συνεργασία, κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Ελπίζω λοιπόν να μπορούμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Και με αυτή την πανέβαση ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψήφιση της εκθέσεως πρόκειται να γίνει το μεσημέρι με τις υπόλοιπες ψηφοφορίες. Πάμε στο επόμενο σημείο σημαντικής διατάξει που είναι η προφορική ερώτηση όσον αφορά τι υπηρεσίε υπηρεσίες που προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή που ασχολείται με θέματα τουρισμού και μεταφορών. Πρώτα-πρώτα, ο εισηγητή για το λόγο, κύριο Μπράιν Σίμψον, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, Μπορώ να μιλήσω εξ ονόματο τη Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Κύριε Πρόεδρε, όσοι παρακολουθούμε τη διαδικασία τη απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, γνωρίζουμε πόσο μακροσκελή είναι αυτή η διαδικασία. Από την αρχή, στη δεκαετία του 1980, το Κοινοβούλιο μα προσπαθεί να διασφαλίσει πω οποιαδήποτε απελευθέρωση δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τι συνθήκε εργασία και θα πρέπει βεβαίω να εγγυάται η καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στου πολίτε η σύγχρονη τεχνολογία αλλάζει δραστικά τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά σε τελική ανάλυση πάντα θέλουν οι άνθρωποι να βλέπουν σε καθημερινή βάση τον ταχυδρόμο τους να τους φέρνει το ταχυδρομείο, την αλληλογραφία. Γι' αυτό λοιπόν η αφετηρία πρέπει να είναι ή ταχυδρομικές υπηρεσίες και όχι μόνο ο ισολογισμός, αλλά και μια κοινωνική υπηρεσία που παρέχεται. Με αυτή την αφετηρία πρέπει να κρίνουμε την οδηγία 2008 κάθετος 6 που θα ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου φέτος. Στόχος της ερώτησης της προφορικής είναι να υπενθυμίσει στην Κομισιόν τις δικλίδες ασφαλείας που έχει θέσει στην οδηγία το Κοινοβούλιο στους τομείς κοινωνικής προστασίας και της παροχής και χρηματοδότησης της καθολικής παροχής υπηρεσίας και να υπενθυμίσει στα καρδιμέλη πως έχουν υποχρέωση να ε, προστατεύσουν αυτά ε, τα πράγματα και όχι όπως έκαναν με την απελευθέρωση των στερεοδρόμων να αγνοήσουν τον νόμο. Και εκεί είναι το δίλημα που αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει υποψία πως η Κομισιόν δεν θα επιβάλλει αυτές τις σημαντικές πτυχές της οδηγίας 2008-6 αλλά με μεγάλο ζήλο θα εφαρμόσει τα της οικονομικής απελευθέρωσης αυτής της οδηγίας και δεύτερον πως τα κράτη-μέλη θα κινηθούν με πάρα πολύ αργό ρυθμό και δεν θα κάνουν τίποτα για να προστατεύσουν τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και δεν θα χρηματοδοτήσουν επαρκώς την καθολική υπαρχή υπηρεσίας. Γι' αυτό υπάρχουν τέσσερα ξεκάθαρα ερωτήματα που απαιτούν τέσσερις ξεκάθαρες απαντήσεις από την Κομισιόν. Και αυτά περιέχονται σε αυτή την προφορική ερώτηση. Δεν θέλουμε τεχνικές απαντήσεις από την Κομισιόν, ούτε να μας πούνε το τι αναφέρουν οι συνθήκες. Τα ξέρουμε αυτά στην Επιτροπή μου. Απαιτούμε εγγυήσει των συμφωνημένων στην Οδηγία 2008 κάθετος 6 ότι θα εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης όλων των εργαζόμενων στον ταχυδρομικό τομέα. Την, απαιτούμε την εγγύηση της καθολικής παροχής υπηρεσία. Θέλουμε να δούμε τις μελέτες που απαιτεί η οδηγία για το κόστος της καθολικής παροχή υπηρεσία ή τουλάχιστον μια ημερομηνία για την ολοκλήρωση των μελετών. Θέλουμε η Κομισιόν να κάνει πλήρη αξιολόγηση αντικτύπου της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς και των αποτελεσμάτων που θα έχει σε όλο τον κλάδο, όχι μόνο στην οικονομική πτυχή. Συνελόντι πιν. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί κάνουμε αυτή την προφορική ερώτηση αυτή τη στιγμή. Δυστυχώ η απάντηση βρίσκεται σε μια υποψία για να μην πω δυσπιστία μετά από χρόνια απελευθέρωσης αυτού του τομέα ότι τα κράτη-μέλη αγνοούν τις κοινωνικές διατάξεις και πως η Κομισιόν τους επιτρέπει να το κάνουν. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί. Εμείς ως Κοινοβούλιο δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνει το ίδιο πράγμα το οποίο συνέβη στους σιδηρόδρομους. Τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει υποχρεώσεις με την οδηγία 2008 κάθος 6 και η Κομισιόν πρέπει να φροντίσει να τις τηρήσουν. Το να μην κάνει κάτι τέτοιο είναι κατά τη γνώμη μας αμέλεια των καθηκόντων της. Ευχαριστούμε, Μπράιον, λέει ο πρόεδρος. Μπράβο, γιατί τελειώσες ακριβώς στα 5 λεπτά. 5-0-0. Μεγάλη επιτυχία. La palabra el comisario señor Barnier para responder a la pregunta en nombre de la Comisión. Και τώρα ο κύριος Μπαρνιέ για να απαντήσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εφτά με οχτώ μήνες είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περίπου. Με ακούσατε πολύ συχνά βέβαια να λέω και τελευταία φορά στις 13 ε, Ιανουαρίου την προσωπική πίστη την οποία έχω την προστασία των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Οι υπηρεσίες αυτές συνδυάζουν την μεγάλη ελεύθερη αγορά από τη μία με τους πολίτες από την άλλη. Ε, θα το πω επίσης αυτό και στην παρουσίαση τον Οκτώβριο του Single Market Act Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την απασχόληση, επιμένοντας όμως ότι δεν θα πρέπει να γνωρίσουμε την κοινωνική και συλλογική διάσταση και εδώ ακριβώς ε, η κοινή ωφέλεια, το καθολικό ε, συμφέρον θα πρέπει να προστατευθούν. Το σχέδιο το οποίο προτείνει ο κύριος Σίμψον έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η προβληματική έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια ε, από την 1η Ιανουαρίου ε, του 2011 ε, σε 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 95 περίπου της 100 του ταχυδρομικού κύκλου εργασιών θα έλεγα θα ανοίξει η αγορά και υπάρχουν τρεις οδηγίες οι οποίες έχουν ουσιαστικά συγκεκριμενοποιήσει τις απόψεις και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένους δημοκρατικούς ελέγχους. Θυμάται ο κύριος Σίμψον, η τελευταία μορφή ελέγχου έγινε το 2008 με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου. 25 χώρες υπερψήφισαν τη μεταρρύθμιση αυτή. Έγινε ανοιχτά με μεγάλη διαφάνεια η μεταρρύθμιση αυτή για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και θα επιτρέψει στον συγκεκριμένο αυτόν τομέα που είναι πολύ σημαντικός 95 δις κύκλος εργασιών, 5 εκατομμύρια έμεσων ή άμεσων θέσεων απασχόλησης. Ο τομέας αυτός λοιπόν θα του επιτρέψουμε να εξελιχθεί, να εξυγχρονιστεί και να ανταποκριθεί με καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες και των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς όταν είναι λελογισμένη και ελεγχόμενη είναι πάντα θα έλεγα εγγύηση για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Λοιπόν, καλύτερες υπηρεσίες και οικονομική ανάπτυξη για καλύτερη ανταπόκριση στους πολίτες. Οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι χρήστες είναι ε, προφανείς λόγω των αλλαγών οικονομικών και κοινωνικών. Έχουμε την τύχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάζουμε εδώ και καιρό τις εξελίξεις του ταχυδρομικού τομέα με προοδευτικό σταδιακό και γαλήνιο τρόπο. Η νομοθεσία πλέον συνοδεύει τις ριζικές αλλαγές στην επικοινωνία, στην ηλεκτρονικοποίηση σε εισαγωγικά της επικοινωνίας και αυτό ε, λαμβάνει υπόψη φυσικά και τις ε, συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης την οποία αυτή τη στιγμή βιώνουμε. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία λοιπόν την οποία συνοδεύσαμε με ηρεμία μέχρι τώρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακοπεί η διαδικασία αυτή για πολλούς λόγους. Καταρχάς η επίτευξη των στόχων της πράσινης βίβλου του 92 εξακολουθεί να είναι θα έλεγα στον συγκεκριμένο τομέα ένας βασικός στόχος οι ε, μεγάλες ταχυδρομικές εταιρείες στην Ευρώπη ξέρουν ε, τι χρειάζεται και έχουν συνεργαστεί μαζί μας για τον καθορισμό των προγραμμάτων. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με τις αρμόδιες κρατικές ρυθμιστικές αρχές. Νομίζω ότι το άνοιγμα στην αγορά γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι οι υπηρεσίες αυτές κοινή ωφέλεια και καθολικού συμφέροντος ε, να παρέχονται με οικονομικό αλλά και υπεύθυνο τρόπο. Νομίζω ότι αν προκαλέσουμε μία διακοπή της διαδικασίας θα προκληθεί μία νομική ανασφάλεια θα έλεγα παράδεκτη αχρίαστη σε αυτή τη φάση και για τους ταχυδρομικούς ε, και για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες και δεν πρέπει απλά ε, να σταθούμε παθητικά στις νέες εξελίξεις. Ακούονται ανησυχίες για την απασχόληση και για τις συνθήκες εργασίας. Γνωρίζω την μεγάλη σημασία που έχουν τα ταχυδρομεία στην απασχόληση και θυμίζω ότι η τρίτη οδηγία δίνει την δυνατότητα στις κρατικές διοικήσεις να μείνουν στα κοινωνικά θέματα και στις κοινωνικές συνέπειες των αλλαγών στον ταχυδρομικό τομέα και οι κοινωνικές συνέπειες θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα σοβαρότατα υπόψη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ανοίγματο των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι προϋποθέσεις ε, να γίνονται σεβαστές. Το 2013 όταν το σύνολο των χωρών θα εφαρμόσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα δημοσιεύσει και μια επίσημη έκθεση αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξουν επιμέρους τομεακές μελέτες και νωρίτερα από το 2013. Νομίζω ότι και αυτά που είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο καλύπτουν τις ανησυχίες σας και έχουμε την πρόθεση, χωρίς να έχουμε την υποχρέωση, να δημιουργήσουμε το 2011 μια ομάδα διαλόγου των χρηστών. Υπάρχει μια ομάδα, όπως ξέρετε, διαλόγου και επαφής των επιχειρήσεων και θα μπορέσουμε έτσι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές, οι μεμονωμένοι πολίτες, τα συνδικάτα, να μπορέσουν γύρω από την ίδια τράπεζα να συζητήσουν το τι συμβαίνει και να μπορούν με τακτόχρον, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα δούμε ποιος θα είναι ο ρυθμός αυτός, να επαληθεύσουμε τη σωστή εφαρμογή των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Αυτές είναι οι εγγυήσεις τις οποίες μπορώ να σας παρέχω και σας υπόσχομαι ότι προσωπικά θα αφιερωθώ στην σωστή λειτουργία αυτής της ομάδας επαφή των Χριστών. Ε. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπή τώρα η σειρά των αγορητών των πολιτικών ομάδων πρώτα-πρώτα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Φέρμπερ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Κύριε Πρόεδρε, ω ηγητή τη ε, Τρίτη Ταχυδρομική Οδηγία χαίρομαι για το ότι συζητάμε σε αυτή τη αυτό το θέμα γιατί είναι σημαντικό νομίζω να δείξουμε το τι έχουμε κάνει και το ότι έχουμε επιτύχει από το 1992 μέχρι σήμερα από την υποβολή της Πράσινης Βίβλου και τα λεπά. Τι έχουμε επιτύχει, η ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι καλύτερη. Θυμάμαι πριν από δύο θητείες λέγαμε πως ε, κατά κανόνα συνηθέστερα έρχεται αυτός ο οποίος έχει πάει διακοπές, επιστρέφει σπίτι του από ότι η κάρτ ποστάλ που στέλνει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ε, έχουμε επιτύχει ποιότητα στον ε, ταχυδρομικό τομέα και εντός των ε, κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η υποχρέωση καθολικής παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ευρώπη και βεβαίως αυτό σημαίνει πως βελτιώθηκε η εκεί που ήταν πάντα καλά μπόρεσε να διατηρηθεί σε αυτό το υψηλό επίπεδο και αυτό νομίζω το εκτιμά και το ανέφερε και ο Επίτροπος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας. Τώρα βεβαίως το θέμα είναι η εφαρμογή της τρίτης οδηγίας και το τι θα γίνει από 1η Πρώτου 2011 που είναι η ημερομηνία της πλήρους απελευθέρωσης οπότε θα πρέπει να διασφαλιστεί η καθολική παροχή υπηρεσίας και θέλω να υπογραμμίσω αυτό το οποίο αναφέρει στην ερώτηση με την σύνδεση που ήταν ε, εκ των ΟΝ ΟΥΚΑΝΕΦ με το ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό το οποίο υπάρχει ως προστασία, ως κοινωνικές προδιαγραφές θα συνεχίσει να ισχύει και μετά την 1η Πρώτου 2011 και οπωσδήποτε θα το προσέξουμε αυτό και δεν θα εξαντληθεί αυτό στη σημερινή προφορική ερώτηση. Πρέπει και η Κομισιόν να δίνει λόγο και θα διαβάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία θα μας πείτε κύριε Επίτροπε και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές για δύο λεπτά ο κύριος Ελχαντραουή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντησή σας και πράγματι νομίζω πως πρέπει να γίνει ένας διάλογος με τους χρήστες που εμείς θεωρούμε ως ομάδα πως είναι απαραίτητος πάντα. Ήμασταν επικριτικοί, γιατί καλό είναι ο στόχο τη αποτελεσματικότητα του κλάδου, αλλά υπάρχουν δύο σημεία κλειδιά για τα οποία θα πρέπει να έχουμε επαρκείς εγγυήσει. Δηλαδή, η κοινωνική πτυχή, οι συνθήκε εργασία και η χρηματοδότηση τη καθολική ε, παροχή υπηρεσία, η οποία θα πρέπει βεβαίω να συνεχίσει να υπάρχει σύμφωνα με την οδηγία. Αυτά συνδέονται μεταξύ του όσον αφορά την κοινωνική πτυχή. Νομίζω πω πλέον το μπαλάκι είναι στα κράτη-μέλη θα πρέπει λοιπόν να, δημιουργηθεί και, να δημιουργηθούν και οι συνθήκε ανταγωνισμού μεταξύ των παλαιών μονοπωλίων και των νέων εταιριών στον τομέα αυτών και αυτό βεβαίω θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το κόστος ε, γιατί το κόστος εργασίας είναι πάνω από το 70% του κόστους του κλάδου οπότε τι γίνεται έχουμε επισφαλείς συμβάσεις και χαμηλούς μισθούς δεν είναι αυτή η Ευρώπη την οποία επιθυμούμε θα πρέπει λοιπόν να πληρώνει το μονοπόλιο, δηλαδή οι μεγάλοι πελάτες, την παροχή καθολικής ε, υπηρεσίας ε, σε αεροκατοικημένες περιοχές. Αυτό ήταν η θεωρία. Στην πράξη, κατ' ουσίαν, το κράτος μέσω επιδοτήσεων θα χρηματοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Και εκεί πέρα βεβαίως ασκείται η πίεση. Εσείς λοιπόν κύριε Επίτροπε θεωρείτε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους οδηγίας, δηλαδή περισσότερη ενταφική και κοινωνική συνοχή. Δεύτερον, Μιλάμε για έκθεση την οποία θα συντάξετε το 2013. Μήπως θα μπορούσατε νωρίτερα να μας πείτε τι γίνεται στα κράτη-μέλη και ειδικά όσον αφορά αυτές τις δύο πτυχές, κοινωνική και καθολική υπηρεσία και τέλος τι θα κάνει η Κομισιόν για να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει να υπάρξουν ίσοι ανταγωνισμού και για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα. Ευχαριστώ. Gracias. Εμείς ευχαριστούμε σαν λέει ο Πρόεδρος και τώρα για τους φιλελευθέρους έχει το λόγο η κυρία Μάισνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζούμε σε μια Ευρώπη όπου θέλουμε πως θα μπορούν, να μπορούν να συνεπάρχουν οι άνθρωποι και να έχουν συνθήκες ζωής που θα είναι καλές και γνωρίζετε πως έχουμε και δημογραφική αλλαγή, δηλαδή έχουμε λιγό, θα έχουμε λιγότερους ανθρώπους που θα ζουν στην Ήπεθρο από ό,τι τώρα. Παρόλα αυτά θέμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τις υπηρεσίες ε, τις οποίες θα είναι και χρειάζονται για να μπορούν να ζήσουν και βεβαίως αυτό συμπεριλαμβάνει και το ταχυδρομείο για να διασφαλιστεί η καθολική παροχή της υπηρεσίας και ακριβώς εδώ πέρα φτάνουμε στο θέμα του πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την παροχή της υπηρεσίας στην Ήπεθρο με λιγότερα λεφτά στο ταμείο και με χαμηλές τιμές και να μπορούμε να πληρώνουμε και τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους με ένα λογικό μισθό. Ε, δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα για τα κράτη-μέλη, το γνωρίζουμε, αλλά αποφασίσαμε και κύριε Επίτροπε αναφέρατε πως ε, αυτό, σε αυτό συμφώνησε και η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών, πως είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε και βλέπω και κάποια δυσκολία εγώ όσον αφορά το να υπάρχει δυνατότητα να κάνουν οι πολίτες τα παραπονά τους, το οποίο αναφέρει η οδηγία και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Ακριβώς γιατί με λιγότερους ανθρώπους θα πρέπει να διατηρηθούν οι υποδομές. Και είπατε κύριε Πρόεδρε πως είστε καινούριος και θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά αντιλαμβάνεστε πως έχουμε ένα σκεπτικισμό στην Επιτροπή μας. Το είπε και ο Μπράιν Σίμψον, γιατί αρμόδια ήταν και για τους σιδηροδρόμους η Κομισιόν για την εφαρμογή και βλέπετε δεν έγινε τίποτα. Και σε άλλους ε, τομείς ε, δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα τα θέλαμε. Το γνωρίζω γιατί το έχουμε και στη Γερμανία αυτό το φαινόμενο. Είναι μια χαρά οι αποφάσεις, ε, συμφωνούμε όλοι και δεν υπάρχει καμία εφαρμογή. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμογιστούν όλα αυτά εδώ πέρα προς συμφέρον των ανθρώπων και των εργαζομένων στα ταχυδρομεία και βεβαίω να το καταφέρετε και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστούμε και τους πλασίνου τώρα για 1,5 λεπτό. Η Ιζαμπέλ Ντιρόν, η αντιπρόεδρο τη ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν αμφισβητώ τη δημοκρατική διαδικασία και τη διαφάνεια που οδήγησε στην υιοθέτηση της οδηγίας αυτής για το άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι θα ήταν εξίσου δημοκρατικό και διαφανές σε μια κάποια φάση να αξιολογήσει κανείς τις επιπτώσεις των εφαρμογών, της εφαρμογής μάλλον αυτών των οδηγιών. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε πολλά κράτη-μέλη και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βελτίωση των υπηρεσιών ή για καλύτερη προσβασιμότητα των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Μιλήσατε για αλληλογισμένη και συνοδευόμενη διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι στην ουσία βλέπουμε να υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση των ιδιωτικών εταιριών, ενώ εμείς θέλαμε να σπάσουμε το κρατικό μονοπόλιο, το αποτέλεσμα λοιπόν δεν είναι αυτό το οποίο όλοι ανέμεναν. Μιλήσατε επίσης για τη συνοδεία της διαδικασίας αυτής και την επίβλεψή της. Πράγματι υπάρχει μια ομάδα ρυθμιστών, αλλά θα ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί το σύστημα στις διάφορες χώρες και στον τομέα της απασχόλησης θα συμφωνήσω με τον Ελ Καντράουι γιατί ξέρω ότι οι νέες θέσεις οι οποίες δημιουργούνται είναι προσωρινές και ανασφαλείς και ο κανόνας είναι η απώλεια των θέσεων απασχόλησης. Ο διάλογος ανάμεσα στους χρήστες είναι σημαντικό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την μεγάλη αγορά με τον πολίτη. Ε, το ταχυδρομείο μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε σε επαφή αυτές τις δύο διαφορετικές ιδέες, αλλά αμφιβάλλω αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό, πρέπει να αξιολογήσουμε ακόμα περισσότερο και με μεγαλύτερη προσοχή και διστακτικότητα την κατάσταση πριν θελήσουμε να αλλάξουμε την ε, κατάσταση ως έχει σήμερα. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε για την Ευρωπαϊκή Ενωτική και για δύο λεπτά και το λόγο κυρίως Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μόλις είπατε πως ε, δηλώσατε όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας πως η εσωτερική αγορά θα αποκτήσει κοινωνικό πρόσωπο και ο καθηγητής ο κύριος Μόντι ε, δίνει το ίδιο βάρος αλλά ζούμε την πραγματικότητα χτες έξω από το κτίριο 100 ταχυδρομικοί διαδήλωσαν μεταξύ των οποίων και ε, ένας Ολλανδός ο οποίος ήταν 55 ετών, έχει δουλέψει μόλις 20 χρόνια στο ταχυδρομείο και αναμένει πως θα απολυθεί. Και θα απολυθούν από ό,τι φαίνεται όλοι οι ταχυδρόμοι ε, στο Ολλανδικό ταχυδρομείο, κάτι το οποίο φαίνεται πως θα οδηγήσει στο να αντικατασταθούν από προσωρινούς εργαζόμενους με πολύ χαμηλότερο εργατικό στόχος και μιλάμε για 50.000 απολύσεις επαγγελματιών, ανθρώπων αξιόπιστων που κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ και δεκαετίες. Γιατί κύριε Επίτροπε ποτέ δεν ερευνήσατε τις κοινωνικές πτυχές της απελευθέρωσης ή μάλλον γιατί δεν είδατε τις μελέτες που υπάρχουν και χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχουν στο peqe.at e και μπορεί να τη διαβάσει ο καθένας. Και βλέπετε τι γίνεται. Κλείνουν, ε, απολύονται άνθρωποι, κλείνουν ε, ταχυδρομεία και η τελευταία ιδέα η οποία αναπτύσσεται είναι να χρειώσουν πολύ ακριβά τους ανθρώπους που ζουν στα βουνά ή στα νησιά για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Γιατί δεν είδατε ποιες είναι οι συνέπειες και για τους ταχυδρόμους και για τους πελάτες και γιατί δεν κάνετε ένα μορατόριο της απελευθέρωσης μέχρι να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης. Αυτό θα πει κοινωνικό πρόσωπο. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπάφτον ε, για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας είναι ο τελευταίος. Πρόεδρε ευχαριστώ. Όταν ζητήθηκε από την Ένωση το άνοιγμα στον ανταγωνισμό για τον κλάδο των ταχυδρομείων τότε κατέστρεψε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί εμείς έχουμε κυρίαρχο κράτος και τα ταχυδρομεία ασχολούνται με, με, με ταχυδρομικές υπηρεσίες και γίνεται ταμιευτήρια και, και πολλά άλλα. Είχαμε 25.000 και τώρα έχουμε τα μισά ταχυδρομεία παρά το ότι έχουν πολύ περισσότερο κόσμο. Και δεν θα ήταν δυνατόν να μείνουν ανοιχτά ταχυδρομεία αν δεν υπήρχε ενίσχυση από το κράτο. Χιλιάδε ταχυδρομεία κλείσανε και έτσι ο κόσμο δεν μπορεί να έχει αυτέ τι υπηρεσίε. Τι πολύτιμε, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο το είχαμε στη Βρετανία. Και ε, ήταν αποτελεσματική η λειτουργία σαν επιχείρηση, ήταν προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο, το αρχιδρομείο Τώρα όμως άνοιξε ο κλάδος και ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και νομίζω ότι είναι ντροπή το ότι δεν μπορούμε να έχουμε ταχυδρομική υπηρεσία ε, μόνο και μόνο για να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία. Τι άλλο θα διαλύσετε αύριο. Θα πρέπει το, το, το Βασίλειο να αποφύγει την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Ευχαριστούμε κύριε Μπάφτον και τώρα Έχουμε τους ε, αγορητές οι οποίοι ε, λαμβάνουν το λόγο για δικό τους λογαριασμό. Ε, πρώτος ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συγχαρητήρια στον κύριο Σίμψον που έθεσε τα σωστά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα αυτή η απελευθέρωση πρέπει να δείξει πως αυτή θα επιτύχει τους στόχους της καλύτερης ποιότητας με καλύτερη τιμή. Γιατί και οι παλαιές κλασικές επιχειρήσεις τα προσέφεραν αυτά. Οπότε θα πρέπει να αποδείξουμε πως με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται κάτι αποτελεσματικότερα. Κατά την άποψή μου νομίζω πως πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά διαφορετικά πράγματα. Το εργατικό δίκαιο παραδείγματος χάρη, οι συνθήκες και οι μισθοί πρέπει να παραμείνουν οι ίδιες. Αυτό θα γίνει μόνο με συλλογικές συμβάσεις και κλαδικές συμβάσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να εμποδίσουμε το κοινωνικό τάμπινγκ. Επίσης, η παροχή καθολικής υπηρεσίας αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές ήδη. Και εδώ πέρα αναμένω λοιπόν από την Κομισιόν μία μελέτη. Κατόπιν κάθε χώρα θα πρέπει να τηρήσει την υποχρέωση να έχει μία ρυθμιστική αρχή ανεξάρτητη για τα ταχυδρομεία που θα πρέπει βεβαίως να λαμβάνει υπόψη και τα παράπονα των καταναλωτών και τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και θα πρέπει να έχει και επαρκές προσωπικό η ίδια. Επίσης, επειδή αυξάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τράπεζες, ασφάλειες, τα πάντα γίνονται μέσω ίντερνετ. Όλα αυτά όμως γίνονται μέσω και των υποδομών του ταχυδρομείου. Αναμένω λοιπόν από την Κομισιόν αξιολόγηση αντικτύπου και για τις κοινωνικές πτυχές. Συγχαίρω την ε, Κομισιόν για τον ε, διάλογο τον ε, κοινωνικό, τον οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μπαρνιέ. Κύριε ευχαριστούμε κύριε κύριε Μπάχ και τώρα 1,5 λεπτό κύριε Τίκαο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο προβλέπεται να γίνει το 2011 τα δε κράτη-μέλη που μπήκαν σε Ευρωπαϊκή το 2004 ε, δίνανται εάν το επιθυμούν να ανοίξουν ε, τον κλάδο στον ταγωνισμό το 2013. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως κλάδος, διότι περισυλλέγει, ε, εξεργάζεται, ε, κάνει τη διαλογή, τη διανομή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, τουλάχιστον πέντε φορές τη βδομάδα τα, τα, τις επιστολές και τα γράμματα ακριβώς όπως προβλέπεται για τις καθολικές υπηρεσίες επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ακόμα και σε μια συγκυρία οικονομική κρίση είναι σημαντικό να μπορούν τα κρατημέλη να έχουν αυτό το δίκτυο υπηρεσιών και να λειτουργεί εύρυθμα ο κλάδο και να μπορεί να υπάρχει ταχυδρομή ακόμα και στην Ήπεθρο. Έχουμε τώρα αυτή την οδηγία η οποία ρυθμίζει την ε, λειτουργία των ταχυδρομείων και ορίζει ποιες είναι οι προβλέψεις που θα πρέπει, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και να πρέπει να, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδοτική κάλυψη για να λειτουργούν καλά τα ταχυδρομεία, να, είναι ε, πανδρομένα όπως πρέπει και να υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις όσον αφορά την απασχόληση, την κατάρτιση και το εισόδημα των υπαλλήλων των ταχυδρομείων. Επομένως είναι σημαντικό μέχρι τέλος του έτους να μας παρουσιάσει η Επιτροπή μία μελέτη που να δείχνει τι επιπτώσεις θα έχει η απελευθέρωση του κλάδου για κάθε κράτος μέλος. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε ε, μια διαφοροποίηση ε, έχοντας δηλαδή και ηλεκτρονικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εσωτερική αγορά και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες υποτίθεται θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2010. Αυτοί που κατοικούν σε γεωργικές περιοχές ε, της Υπέθρου και εκεί είναι και η εκλογική μου περιφέρεια έχουν πάρα πολλές ανησυχίες για την κατάσταση αυτή. Οι ταχυδρόμοι άνδρες και γυναίκες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή των Ιρλανδών στην Ήπεθρο και θα ήθελα να τους τιμήσω για τον εξαιρετικό τους ρόλο και τη μεγάλη σημασία που έχει η παρουσία τους εκεί. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν είναι ένας απλός οικονομικός τομέας, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού των περιοχών της Υπέθρου, ιδιαίτερα και στη χώρα μου όπου το 40% κατοικεί επαναλαμβάνω σε γεωργικές περιοχές. Οι εργαζόμενοι ε, είναι το σημείο επαφής των ηλικιωμένων στην Ήπεθρο με τον υπόλοιπο κόσμο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει έτσι ώστε τα στοιχεία ε, των κοινωνικών ε, παροχών που, παρέχονται, που υπάρχουν μάλλον μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από τις εθνικές αρχές θα πρέπει το ταχυδρομείο να συλλέγεται από παντού και να διανέμεται σε όλες και τις πλέον απόμακρες περιοχές της υπαίθρου όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα με ευχαρίστηση τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομάδα Χριστών, στην οποία θα εμπλέκονται και επιχειρήσεις, συνδικάτα, κοινοβούλια και κυρίως οι απλοί χρήστες. Είχαμε δεχθεί πρόσφατα μια αντιπροσωπεία των εργαζομένων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες εδώ και λίγα χρόνια και έχουμε την υποχρέωση να τους εκπροσωπήσουμε σωστά και να εκπροσωπήσουμε φυσικά και τις ανάγκες τις οποίες καλύπτουν, ανάγκες κοινή ωφέλεια, ανάγκες καθολικού συμφέροντος, ε, που πάντα υπήρχαν εδώ και αιώνες στο σύνολο των χωρών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίχτενμπέργκερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να σας πω πως από τις βελτιώσεις που μας υπόσχονται μέσω της απελευθέρωσης δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχω δει πάρα πολλά. Αντιθέτως, αυτό το οποίο λαμβάνουμε εμείς ως βουλευτές ως μήνυμα είναι η επιδίνωση. Μειώνονται οι υπηρεσίες στην Ήπεθρο ήδη σήμερα. Η πρόσβαση στα χειδρομικές υπηρεσίες στην Ήπεθρο πλέον δεν είναι εγγυημένη, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν δύσβατε οικισμοί. Περισσότερες θέσεις εργασίας, ναι, αλλά είναι μίνι θέσεις εργασίας, από τις οποίες δεν μπορεί να ζήσει κανείς είναι ένα βοήθημα αν θέλετε για μια οικογένεια. Αν δούμε λοιπόν θεωρούμε χρήστες μόνο την διαφήμιση αυτοί ναι έχουν όφελος γιατί οπωσδήποτε α, αυτόν ο τζίρος βελτιώθηκε η καθολική παροχή υπηρεσίας τώρα φαίνεται πώς θα πρέπει να πληρωθεί από τα κράτη-μέλη τα οποία είναι υπό τεράστια πίεση γιατί βεβαίως ο προϋπολογισμός είναι πλέον υποπίεση και θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι επιδοτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση κύριε Επίτροπε θα έπρεπε νομίζω να δούμε τι γίνεται, για να κάνετε και μια αξιολόγηση αντικτύπου, για να δείτε πως υπάρχει επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιδείνωση κατά των οχυδρομικών. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό η κυρία Ζαμπίνε Βίλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο επίπεδα έχουμε στην απελευθέρωση που εφαρμόζονται ήδη. Η Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιεύσει κάποια δική της μελέτη που να ασχολείται μόνο με τις κοινωνικές πτυχές και τις συνέπειες απελευθέρωσης της αγοράς στον ταχυδρομικό τομέα. Κύριε Μπαρνιέ, σας ερωτώ, πότε θα μας δώσετε επιτέλους στο Κοινοβούλιο αυτή τη μελέτη. Χτες ακούσαμε διαφόρους υπαλλήλου των ταχυδρομείων από διάφορα κράτη-μέλη πως πλέον απολύονται μαζικά και επαναπροσλαμβάνονται με χειρότερες συνθήκες. Η πολιτική του ανταγωνισμού δεν μπορεί να γίνεται στις πλάτες των εργαζομένων. Εάν η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θέλουν να κάνουν κάτι για τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει η τρίτη φάση της απελευθέρωσης να μην λάβει χώρα. Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και η ποιότητα της καθολικής παροχής υπηρεσιών πρέπει να ερευνηθούν σοβαρά. Απαιτούμε λοιπόν με εφαρμογή της τρίτη φάση απελευθέρωση των ταχυδρομείων για του πελάτε και για του εργαζόμενου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. 1,5 λεπτό η κυρία Τούν Ουντ Ευχαριστώ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι συζητάμε μια σημαντική απόφαση προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αυτή είναι η οδηγία για την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες κοινότητας. Πρέπει όμως να φροντίσουμε για την ε, σωστή εφαρμογή ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά τα οποία είπατε κύριε Επίτροπε, προκύπτει πώς θέλετε να συνεργαστείτε με όλα τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι για το ότι η ομάδα αυτή ξεκίνησε τα της ρύθμισης αυτομέα. Ελπίζω λοιπόν να μπορεί να υπάρξει εδώ πέρα κάποια εξυγίανση. Το άνοιγμα των αγορών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και βλέπω πως υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, λύσεις της Κομισιόν απέναντι στο πώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν δραστηριότητε τους οι ανεξάρτητες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι παρατηρείται και την εφαρμογή, αλλά υπάρχει και άλλο ένα θέμα. Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα αν θέλετε χρειάζεται κάποια σύμβολα είναι ο ύμνος, η σημαία το νόμισμα αλλά ο, οπωσδήποτε και μια κοινή αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών νομίζω καλό είναι και αυτό ένα λεπτό για την παρέμβαση η κυρία Σαρακιάνη παρακαλώ η ολοκλήρωση τη εταιρική αγορά στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών μέχρι το τέλο του χρόνου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Θα ήταν όμω σωστό η Επιτροπή να προβεί σε μια αξιολόγηση επίπτωση και αντίκτυπου, όπω ανέφεραν άλλωστε ορισμένοι άλλοι συνάδελφοι, όσον αφορά το άνοιγμα τη αγορά στον τομέα αυτό. Ακριβώ για να καταλάβουμε καλύτερα τι χρειάζονται οι πολίτε. Πώ ε, ε, προτίθεται να διασφαλίσει την προστασία ε, του συμφέροντο των πολιτών που ζουν σε δύσβατε περιοχέ, όπω για παράδειγμα οι ορεινέ περιοχέ έτσι ώστε να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν τακτικά το ταχυδρομείο και τα γράμματά του. Και ποια μέτρα προτίθεται να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι ε, αυτή η οδηγία ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να, ε, για να μα οδηγήσει στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία και έχουν όλα τα μέσα για να το πράξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό ε, έχει το λόγο η κυρία Ισαΐα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε το άνοιγμα των υπηρεσιών των ταχυδρομείων για τον ανταγωνισμό δημιουργεί ανησυχίες σε πολλά κράτη-μέλη για την περαιτέρω διαθεσιμότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε μια μεγάλη χώρα όσον αφορά το εμβαδόν της όπως είναι η Φινλανδία και που είναι αραιοκατοικημένη υπάρχει ο φόβος ότι μόνο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές θα υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες και όχι στις κερδοφόρες αραιοκατοικημένες περιοχές. Εκεί το κόστος θα το πληρώνει το σύνολο. Έτσι λοιπόν τέσσερις φορές είναι ακριβότερη και πολλές φορές και σε κάποιες, σε κάποιες περιοχές δέκα φορές ακριβότερες οι υπηρεσίες αυτές σε αραιοκατοικημένες περιοχές από τις επικνοκατοικημένες περιοχές. Πρέπει να διασφαλίσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Θα ήθελα να μας πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα διαμορφωθεί ο ανταγωνισμός και πώς θα είναι αυθεντικός και γνήσιος όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών όταν βλέπουμε ότι για κάποιους παρόχους υπηρεσιών είναι πολύ αυστηρότερες οι διατάξεις από ότι για κάτι άλλους. Κυρίως ε, πώς το κόστος των συνολικών αυτών ε, ε, κοινοφελών υπηρεσιών θα καλύπτεται. Υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Η πιο απλή είναι να ε, καλύπτονται με έξοδα των φορολογουμένων οι μη κερδοφόρες αυτές οι υπηρεσίες. Στη Φιλανδία θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε μια παράλογη κατάσταση. Βλέπουμε ότι σε σχέση με το κέρδος του κρατικού οργανισμού είναι 100 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Όμως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε δαπάνες εξίσου υψηλές από το προϋπολογισμό προκειμένου να μπορούν να σημειώνουν κάποιες επιχειρήσεις μεγάλα κέρδη στις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Το ερώτημα λοιπόν είναι η οδηγία αυτή δίνει την δυνατότητα να υπάρχει ένα τέλος που θα εισπράτεται για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ώστε να μπορούν να καλύπτονται οι υπηρεσίες αυτές και στις άρεο κατοικημένες περιοχές. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Φερνάντε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε είναι ένα θεμελιώδε μέσο επικοινωνία. Διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στον ανταγωνισμό και στην ανταγωνιστικότητα και στου στόχου τη κοινωνική συνοχή, οικονομική συνοχή και συνοχή των μερών τη επικράτειας. Έτσι δεν είναι δυνατόν να μην έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι υπηρεσίε οι κάτοικοι τη υπαίθρου στο ίδιο επίπεδο υψηλών υπηρεσιών. Οι πιο απομονωμένε περιοχέ έχουν δικαίωμα να έχουν αναβαθμισμένε υψηλή ποιότητα ταχυδρομικέ υπηρεσίε. Βλέπουμε ότι στα κράτη-μέλη, όπω είναι η περίπτωση τη Πορτογαλία, υπάρχει μια μείωση των σημείων πρόσβαση σε αυτέ τι υπηρεσίε στον χώρο τη υπαίθρου και υπάρχει επιδείνωση τη ε, ποιότητα. Η ποιότητα πρέπει να αναβαθμιστεί και να διατηρηθεί, αλλά ποτέ να επιδεινωθεί ή να μειωθεί. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχουμε αρνητικέ επιπτώσει όσον αφορά του όρου εργασία και του όρου μισθοδοσία των εργαζομένων στα ταχυδρομεία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε οι ανταγωνιζόμενοι όσον αφορά υπηρεσίε, μόνο να θέλουν να πάρουν το φιλέτο αφήνοντα τα κόκαλα για του άλλου. Εξηγώ τι εννοώ. Αναφέρομαι για παράδειγμα στου ανταγωνιστέ που θέλουν υποτίθεται να παρέχουν υπηρεσίε, μόνο όμω, εκεί όπου η διανομή είναι κερδοφόρα ή με άλλα λόγια στις ζώνες με μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμιακή. Έτσι απαιτείται η με αλλα λογια στι ζωνε με μεγαλυτερη Επιτροπή να βρει λύσει να βρει λύσει για να αποφύγουμε τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα. Να μην ανακύπτουν αυτά τα προβλήματα. Και έτσι θα πρέπει η αντίστοιχη νομοθεσία να είναι σεβαστή και να τηρείται. Και πρέπει, αν είναι αναγκαίο, να βελτιωθεί κιόλα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, η τελευταία παρέμβαση σε αυτό το γύρο θα είναι για 1,5 λεπτό τη κυρία Σοφιοκόνη. Παρακαλώ. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Στι σύγχρονε κοινωνίε, οι υπηρεσίε αποτελεσματική επικοινωνία είναι ουσιώδει τόσο για, την, για τις ίδιες επιχειρήσεις αλλά και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την άποψή μου αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για αυτό τον τομέα δραστηριοτήτων και μάλιστα την εποχή όπου η τεχνολογική εξέλιξη και η οικονομική κρίση ε, ε, κατέστησαν ιδιαίτερα ευάλωτους τους παραδοσιακούς μεταφορείς. πιστεύω ιδιαίτερα στην κοινωνική και οικονομική συνοχή, στην εδαφική συνοχή, στην οποία ε, σε τελευταία ανάλυση εντάσσονται και αυτές οι υπηρεσίες. Ω πρόεδρο τη Μικτή Επιτροπή για τι ε, Δημόσιε Υπηρεσίε, ε, ε, πιστεύω ότι όσον αφορά αυτέ τι υπηρεσίε γενικού οικονομικού συμφέροντο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και μην ξεχνάμε τη διαδήλωση χθε στο Στρασβούργο των υπαλλήλων τεχνικών υπηρεσιών. Γι' αυτό η απελευθέρωση θα πρέπει να γίνει ει βάρο των συνθηκών εργασία των εργαζομένων και τη ποιότητα των υπηρεσιών. Η Οδηγία 2008 εξασφαλίζει την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών αλλά γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο, κυρίω όσον αφορά τι υποχρεώσει σε θέματα καθολικών υπηρεσιών. Επίση, να σα πω ότι οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να εξελιχθούν διαφοροποιώντα τι δραστηριότητέ του και με αυτόν τον τρόπο του οδηγήσουν και σε περισσότερα έσοδα. Ε, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επαγρυπνεί και να εξασφαλίσει ε, πολύ αυστηρή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα αυτό θα πρέπει να υπάρξει ε, μία μείζον διαρθρωτική αναδιάρθρωση ε, στον τομέα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ε, και τις απαιτήσει της οικονομικής εποπτείας. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στι ε, παρεμβάσει των Catch the Eye. Έχουμε πολύ περισσότερου ε, ε, συναδέλφου που θέλουν το λόγο, αλλά θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε μία προσπάθεια να δώσουμε σε όλου το λόγο. Αν όμω ακολουθήσετε αυστηρά το όριο του ενό λεπτού. Θα σας, είμαι αναγκασμένος να σας διακόψω μόλις περάσει το ένα λεπτό. Κύριος Νικολάς είναι ο πρώτος ε, ομιλητής. Um, Σα ευχαριστώ πολύ. Το Δεκέμβριο 2010 είχαμε ένα σημαντικό ορόσημο που σημειώθηκε στην υλοποίηση και ολοκλήρωση τη κοινή εσωτερική ενιαία εσωτερική αγορά για ταχυδρομικέ υπηρεσίε. Άρχισε και άνοιξε τότε το άνοιγμα τη αγορά για όλου του παρόχου και ο ανταγωνισμό ενισχύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί καινοτομίε σε αυτό το τομέα και μάλιστα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και αυτό το θεωρώ σημαντικό. Το θεωρώ σημαντικό διότι η μονοπωλιακή οργάνωση των εθνικών αγορών έχει πολύ έντονο μονοπωλιακό ακριβώ χαρακτήρα και αυτό οδηγεί στο να αυξάνουν οι τιμέ και αυτό έχει αρνητικέ επιπτώσει επί των καταναλωτών. Υποστηρίζω την, απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση των, ε, ε, των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αυτό θα οδηγήσει στην κατάργηση των μονοπωλίων, θα βελτιώσει τις τιμές και θα είναι προς όφελος των καταναλωτών οπωσδήποτε και δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζομένους. Ο Ταραμπέλα στη συνέχεια παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, και εγώ είχα ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο ποιε θα ήταν οι αρνητικέ επιπτώσει τη απελευθέρωση αυτή από τη στιγμή που πάρα πολλέ έρευνε έχουν δείξει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλε δυσλειτουργίε, αυξάνονται οι τιμέ, μειώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών και εξαφανίζεται η διαφάνεια. Η Επιτροπή έχει αναλύσει την απελευθέρωση τη αγορά ηλεκτρική ανέργεια στι αρχέ του 2010, αλλά θα πρέπει να αναλύσει και την, το ενδεχόμενο απελευθέρωση και στι ταχυδρομικέ υπηρεσίε, λαμβάνοντα υπόψη ε, την ανάγκη για υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. Έχει έλθει λοιπόν πλέον η ώρα να είμαστε αντικειμενικοί, να εμβαθύνουμε στο θέμα και να μην διαπράξουμε τα λάθη που έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν σε απελευθερώσεις άλλων κλάδων της οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τον διάλογο και θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Περιμένουμε πολύ περισσότερα από εσά, ε, κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει προς τα εμπρός. Ευχαριστώ κύριε Τραβέλο, λόγο στην κυρία Χάρκιν. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν την οδηγία με αρκετό περιθώριο ελιγμών ούτως ώστε να, να πληρούν τις προϋποθέσεις για την προστασία των εργασομένων. Εμείς ζητήσαμε αξιοπρεπή απασχόληση στην διαδήλωση και η αξιοπρεπής απασχόληση ουσιαστικά χάνεται και αντικαθίσταται από αβέβαιη και προσωρινή εργασία. Οι πολίτες ανησυχούν, αλλά και οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι ανησυχούν για την απώλεια θέσεων απασχόλησης και ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ανησυχίες αυτές. Εκπροσωπώ μια ε, περιφέρεια η οποία ανησυχεί ιδιαιτέρως για τη διασφάλιση της ε, ποιότητας των υπηρεσιών και η οποία επιθυμεί τη διατήρηση της ε, ταχυδρομικής υπηρεσίας πέντε μέρες την εβδομάδα. Όντως χρειάζεται μορατόριο ως προς την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Διακόπτει ο Πρόεδρος, ο κύριος Φεραίρα έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, σε όλη την Ευρώπη είμαστε μάρτυρες από πλευρά των πληθυσμών και των εργαζομένων σε μια πραγματικότητα. Η απελευθέρωση των υπηρεσιών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το αντίθετο από ό,τι δηλώθηκε αρχικά και από ό,τι είχε παρουσιαστεί, οδήγησε σε μια σημαντική επιδείνωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και σε μια επίθεση χωρί προηγούμενο στα δικαιώματα των εργαζομένων αυτού του τομέα. Όπω και σε άλλου τομεί, η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση οδηγεί σε επικέντρωση μονοπωλιακή σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι συνέπειε είναι ορατέ, Ακόμα και σε χώρε όπου βρίσκεται αυτή η διαδικασία σε πιο αποθυμένη ε, φάση. Και πρέπει να πούμε ότι η διανομή σε σχέση και με την ε, διαμόρφωση των τιμών και το κοινωνικό dumping, για αυτού του λόγου ε, ενώνονται σε ένα κοινό αγώνα οι εργαζόμενοι κατά τη ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Θέλουμε να δώσουμε αξία σε αυτόν τον αγώνα και να σημειώσουμε την αξία αυτών των μαχών. Και θα πρέπει να λάβει η Επιτροπή αυτά υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φερέρα. Η κυρία Ελίν Ρέγνερ παρακαλώ έχει τον λόγο. Κύριε Επίτροπε, μόλις ε, στη συζήτηση για τις ε, καλύτερες, ε, την διαμόρφωση καλύτερων συνθήκων εργασία είχα συμμετάσχει. Και αυτό δείχνει ότι δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιπτώσεις αν προηγούμενα είχαμε την καλύτερη διαδικασία, την νομική διαδικασία και μια πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δημοσίευσε καμιά μελέτη που να ασχολείται με τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις συνέπειες ε, της απελευθέρωσης των ταχυδρομείων. Η Επιτροπή υποστηρίζει μόνο τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ε, ώστε να, να υπάρξει ένας ανταγωνισμός ε, χωρίς όρια. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν χαμηλόμιστοι και όχι και με ιδιαίτερα προσόντα εργαζόμενοι. Και βλέπουμε ότι έχουμε και διαφορετικέ τιμέ για διαφορετικέ περιοχέ. Γι' αυτό ερώτηση προ εμά, κύριε Επίτροπε. Δεν ματώνει η καρδιά σα όταν βλέπετε ότι ενάντια στην θέληση των εργαζομένων και των συνδικάτων τα ταχυδρομεία στη Γαλλία ιδιωτικοποιούνται. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ κύριε Ρίτνερ. Στη συνέχεια η κυρία Ινέσα Γιάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σε χώρε όπου έχει ήδη λάβει χώρα η απελευθέρωση, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία κτλ, έχει ήδη φανεί ε, ότι δεν δίνεται εναλλακτική λύση στους εργαζόμενους και ούτε πάνε καλά οι επιχειρήσεις αυτές. Θα πρέπει να εγγυηθούμε τις καθολικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια στην ίδια τιμή και ε, τουλάχιστον πέντε μέρες την εβδομάδα. Κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την υποβάθμιση ή μη της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης για να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping και να εφαρμόσουμε σωστά την νομοθεσία όπως το απαιτεί το Κοινοβούλιο. Τη διακόπτει ο Πρόεδρος, την κυρία Αγιάλα. Ήθελα να μείνω στο ένα λεπτό. Γι' αυτό μιλούσα γρήγορα κύριε Πρόεδρε. Λέλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ και θα πρέπει ο κύριος Μπαρνιέ να μας δείξει ότι όντως η οδηγία θα κινηθεί προς ε, την κατεύθυνση των επιθυμιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση ως προς τα σημεία πρόσβασης και θα πρέπει ε, να υπάρχουν ε, δικαιώματα διεκδίκησης και αναφοράς. Ο κύριος Μπιδήλο έχει το λόγο. <clears throat> Ε, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κύριε Μπαρνιέ, το πέρασμα από, τη διαχείριση εκ μέρους των εθνικών κρατών σε μια διαχείριση εκ μέρους της ολόκληρης της Ευρώπης ε, είναι ε, κάτι το σημαντικό και εγώ συμφωνώ βεβαίως. Αλλά ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί επαρκώς το θέμα του κόστους καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή διανομή, θα πρέπει να υπάρχει σωστή διανομή των, του ταχυδρομείου λαμβάνοντας υπόψη τις δύσβατες περιοχές, τις απομακρυσμένες περιοχές, το θέμα της διασύνδεσης των διαφόρων χωρών και των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση ε, της σταθερής απασχόλησης ε, και όχι της απασχόλησης σε προσωρινή βάση. Το κόστος ε, ε, των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Τελείωσε ο χρόνος, τον διάκοψε ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Ε, ε, με, με εντυπωσιάζει ο κανονισμό και το γεγονό ότι ε, ε ο υποβάλλον την επερώτηση δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο για να απαντήσει. Άρα λοιπόν ο κύριο Σίμψον ε, θα πρέπει να προσφύγει στη διαδικασία catch the eye για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Ενώ εγώ νομίζω θα μπορούσε να του έχει δοθεί περισσότερο χρόνο. Κύριε Σίμψον, στα πλαίσια των, της διακριτικής ευχέρειας που έχω ως πρόεδρος, θα σας δώσω δύο λεπτά για να μπορέσετε να απαντήσετε σε όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν γιατί είστε ε, εσείς που υποβάλλετε την ερώτηση. Παρόλο που παίρνετε το λόγο τυπικά στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το γεγονό ότι πάρα πολλοί ε, ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία ε, Catch the Eye δείχνει ακριβώ το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, επιτρέψτε μου να τονίσω ε, αυτό το γεγονό και στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Άκουσα την απάντηση του Επιτρόπου και ε, από πολλέ πτυχέ ε, με ικανοποίησαν αυτά τα οποία άκουσα. Αλλά πρέπει να σα πω ότι υπάρχει βαθύτατη ανησυχία στο Κοινοβούλιο για το γεγονό ότι με την απελευθέρωση των χειδρομικών υπηρεσιών οι κοινωνικέ συνθήκε, οι συνθήκε εργασία των εργαζομένων, καθώ επίση και αυτέ καθεαυτέ οι υπηρεσίε όπω εμπεριέχονται στα πλαίσια των καθολικών υπηρεσιών, θα απο αποδυναμωθούν στο βωμό της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα αυτό και ελπίζω στην απάντησή του ο Επίτροπος να τοποθετηθεί. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να θίξω ε, αφορά αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της ομάδας EFD ε, Ευρώπη και Δημοκρατία ε, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και με το γεγονό ότι έκλεισαν κάποιες ταχυδρομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ως απόρρια της απελευθέρωσης. Κοιτάξτε, θα πρέπει να το δούμε το σημείο αυτό με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο. Το κλείσιμο ορισμένων ταχυδρομείων στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν απόφαση της χώρας αυτής. Ήταν μια απόφαση ε, που οφείλεται στο γεγονός ότι μείωσε τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις η κυβέρνηση προς τα ταχυδρομεία και ε, άλλαξε ε, τη μέθοδο πληρωμής. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, υπήρξαν κάποιες, ε, ε μείωση δηλαδή των επιχορηγήσεων προς, το, προς τα βασιλικά ταχυδρομεία, αποτέλεσμα να κλείσουν κάποια ταχυδρομεία. Το θέμα του opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πραγματικά ένα από τα πιο αστεία πράγματα που έχω ακούσει στη ζωή μου όσον αφορά τα ταχυδρομεία. Ακόμα και ο ε, πιο φανατικός υπέρ της απελευθέρωσης ε, ε μάλλον οι κυβερνήσει της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από τη Θάτσερ στον Τζον Μέιτζορ στον Μπλερ ήταν όλοι υπέρ τη απελευθέρωση. Ε, μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν χεσμολά όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έληξε ο χρόνος σας. Θα τελειώσουμε λοιπόν τη συζήτηση με την αντίδραση του ε, κυρίου Επιτρόπου, του κυρίου Μπαρνιέ. Ε, υπήρξαν πολλές ε, παρεμβάσεις και ε, παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν σε διάφορα ζητήματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Κύριε Σίμψον, σας ευχαριστώ που θέσατε το θέμα αυτό που πυροδότησε την έναρξη της συζήτησης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο-τρία πράγματα ε, πριν ε, μπω στον πυρήνα της απάντησης που θα δώσω. Όπως είπα προηγουμένως, αλλά και όπως όλοι αντικειμενικά αναγνωρίζουν, αυτή η ελεγχόμενη, αυτό το ελεγχόμενο άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν έγινε ούτε λάθρα, ούτε κρυφά, ούτε πολύ γρήγορα, ούτε τυχαία. Έγινε με μια ε, τακτική ε, διαδικασία δημοκρατικής ε, πιστοποίησης, αν θέλετε, και κατοχήριωσης και ο κύριος Μάρκος Φέρπερ και εσείς κύριοι Σίμψον και πολλοί άλλοι ήσασταν μέτοχοι αυτής ε, της διαδικασίας εξ αρχής. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο που έχουμε φτάσει. Είχαμε μια προοδευτική ε, κίνηση, τίποτα δεν έγινε βιαστικά και τίποτα δεν έγινε κρυφά και μυστικά. Και Καθόλου δεν θέλουμε να προδικάσουμε ε, τα πράγματα, ούτε να κινηθούμε εμείς ως Επιτροπή γρηγορότερα από ό,τι απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, γνωρίζω πολύ καλά τι προβλέπουν οι συνθήκες και τι, έχουν, ε, τι έχει διατυπωθεί στα κείμενα. Εγώ προσωπικά έχω παλέψει πάρα πολύ, ε, ήμουν Ευρωπαίος Επίτροπος όταν συζητεί το η συνθήκη της Λισαβόνας και τα διάφορα θεσμικά θέματα τότε και οι διάφορες θεσμικές μεταρρυθμίσεις τότε και εγώ είχα πραγματικά διεξάγει ένα πολύ σημαντικό αγώνα υπέρ της συμπερίληψης του όρου εδαφική συνοχή και κοινωνική συνοχή. Και βεβαίως περιλαμβάνουμε εκεί το δημόσιο τομέα, τις δημόσιες υπηρεσίες δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη ουσιαστικά συνίσταται σε μια μεγάλη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη αγορά. Είναι ένας κοινό χώρος διαβίωσης οικονομικής, κοινωνικής και ανθρώπινης, αν θέλετε, συμβίωσης και ζωής. Αυτές ήταν ανέκαθεν οι αρχές μου, οι πεπιθήσεις μου και Αυτές τις αρχές υπερασπίζομαι καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου και θα συνεχίσω βεβαίως να το κάνω καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας μου ως επιτρόπου. Από εκεί και πέρα. Έχουμε και το κείμενο αυτό καθεαυτό της οδηγίας για την απελευθέρωση των ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δεν πιστεύω ότι ένα μορατόριο ή εν πάση περιπτώσει μια έτσι βίαιη τροχοπέδη ή παρεμπόδιση της εφαρμογής της οδηγίας θα ήταν χρήσιμη. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν εις βάρος των επιχειρήσεων αλλά και του ε, χρήστη, του καταναλωτή των υπηρεσιών αυτών. Τούτων λεχθέντων θα εκτεληχθεί όλη αυτή η διαδικασία και καθώς ο χρόνο θα εξελίσσεται, εμείς οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε και να επαληθεύσουμε ότι ε, θα εξελίσσεται σύμφωνα πάντοτε με τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Έχουμε λοιπόν την καθολικότητα των υπηρεσιών αυτών, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, και είναι κάτι το οποίο κατοχυρώνεται στο κείμενο της οδηγίας. Διάφορους μηχανισμούς έχουμε στη διάθεσή μας για να επαληθεύσουμε του λόγου του αληθές και στην περίπτωση των ε, δημοσίων προμηθειών αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Διασφαλίζονται λοιπόν όλα αυτά. Ε, έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο ως απαραίτητη προϋπόθεση ημέριντα για τις συνθήκες εργασίας. Κοινωνική προστασία λοιπόν. Το λέω για να ε, απαντήσω στην κυρία Τζιγόν και σε άλλους καθίσταται σαφές το κείμενο ότι τα κράτη-μέλη ε, θα διαθέτουν μέσα στη διάθεσή τους στο πλαίσιο της, ε, του εργατικού δικαίου, της εργασιακής νομοθεσίας που έχουν υιοθετήσει για να αποφευθούν πρακτικές τύπου κοινωνικού dumping. Και ότι θα έχουν τα κράτη-μέλη τη σωστή προσέγγιση ε, για την προστασία των θέσεων απασχόλησης. Μπορώ να σας δώσω αυτά αλλά και πολλά περισσότερα παραδείγματα της διατύπωσης του κειμένου, παραδείγματα τα οποία ουσιαστικά αποτελούν δικλείδες ασφαλείας και για τα κράτη-μέλη και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για εσάς μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίως τα μέλη του Συμβουλίου. Και εγώ ήμουν ερετός ερετός ε, για πάνω από 20 χρόνια και ε, μάλιστα σε μια εξαιρετικά ορεινή περιοχή και γνωρίζω πολύ καλά τις ανάγκες ε, για την ταχυδρομική εξυπηρέτηση των κατοίκων και των περιεχών αυτών. Έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία λοιπόν για την, ως προς την Ήπεθρο και ως προς τις αγροτικές περιοχές. Θέλω να σας υπενθυμίσω το εξής. Εάν τα κράτη-μέλη δεν σεβαστούν τουλάχιστον ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις, τότε θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, έχει μέσα στη διάθεσή της για να δράσει προς όφελος των πολύ ορεινών ή των πολύ αγροτικών ε, και απομακρυσμένων περιοχών. Πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, χωρίς όμως να βιαστούμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα διατυπωθέντα στο κείμενο γίνονται σεβαστά. Βεβαίως θα πρέπει να εκπονούνται μελέτες ε, που να προτείνουν διορθωτικές κινήσεις εάν αυτό χρειαστεί. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στις πρώτες μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί, κάτι το οποίο και εγώ σας επιβεβαιώνω και όντω φέτος θα εκπονήσουμε μια πρώτη μελέτη, έχει ήδη ξεκινήσει η σύνταξή της, όπου θα συμπεριληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και η μελέτη αυτή θα ασχοληθεί και με τις πιο πρόσφατες τάσεις σε θέματα απασχόλησης. Έχουμε επίσης μελέτη επίσημης αξιολόγησης, επίσημη έκθεση που θα πρέπει να υποβάλουμε υπόψη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, το 2013 μετά την πλήρη απελευθέρωση και υπάρχει και ο διάλογος μεταξύ των χρηστών, ε, στον οποίο συμμετέχετε και εσείς, χρήστες δηλαδή τα συνδικάτα, οι επιχειρήσεις αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες, οι πολίτες. Θα εξεταστούν λοιπόν οι μελέτες αξιολόγησης που θα υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου. Να απαντήσω λοιπόν στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να πω το εξής. Προσδίδω ιδιαίτερη σημασία τόσο όσο και εσείς στη σωστή εφαρμογή της οδηγίας αυτής δεν θα πρέπει να επιβαρύνει ή να αποβεί εις βάρος των πολιτών και των χρηστών των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα, την ακρίβεια και την εντιμότητα στα λεχθέντα στα περιεχόμενα των διαφόρων μελετών αξιολόγησης που έχουν εκπονηθεί ή που θα εκπονηθούν. Η συζήτηση που κάνουμε και που θα κάνουμε για την ύπαρξη αυτών των μελετών είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να μην αδικούν οι διάφορες μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αποφάσεις που έχουμε εμείς λάβει όλοι από κοινού. Όταν γίνεται λόγος για θέσεις απασχόλησης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, για κοινωνική προστασία, για εδαφική συνοχή, για ποιότητα στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, να πούμε ε, πόσα οφείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πόσα μπορεί να οφείλουμε ε, αλλού, ποιος έχει αρμοδιότητα γιατί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για ποιο πράγμα έχει αρμοδιότητα, οι κυβερνήσεις για ποιο πράγμα αντιστοίχω οι επιχειρήσεις και ούτω Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και θα ήθελα να πω ότι θα παρακολουθήσω εκ του σύνεγγυς την ε, θεσμοθέτηση της ομάδας ε, διαλόγου μεταξύ των χρηστών για να αποδείξουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή την βούλησή μας πραγματικά ε, να ρυθμίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό τον κλάδο της αγοράς, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Σε 8 λεπτά θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες, επομένως αναστέλουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για λίγα λεπτά ε, μέχρι την έναρξη των ψηφοφοριών. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο της ημέρας.